Θα και πάλι γιατί καθερίσαμε με τη συζήτηση για την Κουβά. Σαλαφράγκα, άντρη και Προσπαθήστε παρακαλώ λίγο να συνεργαστούμε. Η συζήτηση γίνεται σε μια στιγμή κλειδί επειδή αυτή τη χρονιά ήμασταν όλοι μάρτυρες ε, πολύ ε, μεγάλων αλλαγών στις σχέσεις με την Κούβα. Είναι Κύριε σημασία συζήτηση. Το Κοινοβούλιο προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εξέλιξη των σχέσεων με την Κούβα. Αυτό φαίνεται επίσης από το ότι συνδιοργανώνουμε τη διάσκεψη με τη Eurolat. Καλωσορίζω τον πρόεδρό της, κύριο Αντώντο. Στις 6 Ιουνίου έγινε συζήτηση στα πλαίσια του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αβάνα. Πρώτη φορά οργανώταν τέτοια συνεδρίαση στην Κούβα. Η διμερή συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας με την Κάβα, ε, Κούβα συγγνώμη, ε, υπογράφηκε στις 6 Ιουνίου. Είναι δημόσιο το έγγραφο, έχετε αντίτυπο στον ηλεκτρονικό σας φάκελο. Το Κοινοβούλιο του επόμενου μήνε θα εξετάσει το περιεχόμενο της συμφωνίας που σηματοδοτεί ε, αρχή νέας εποχή στις σχέσεις με την Κούβα και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πάγωσαν οι σχέσεις με τη ΣΥΠΑ φέτος, ε, ξεπάγωσαν μετά, έγινε η επίσκεψη Ομπάμα. Ε, το γραφείο Ζαχάροφ κατήγγειλε την κατάσταση των ακτιβιστών και αναφέρει ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση τον τελευταίο χρόνο. Ο κ. Γιγέρμο ε, Φαρίνιας, που ήταν υποψήφιος για το Βραφείο Ζαχάροφ το 2010, είναι ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζει στην Κούβα και ε, έχει ενεργό ρόλο και στο Κοινοβούλιο σε σχέση με το βραβείο Ζαχάροφ. Ε, έκανε απεργία πείνα αρχές του 2016. Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας. Ο κύριος Αλεχάνδρο Γκονζάλε Ράγα είναι επίση μαζί μας και πέρα από τον κύριο Φαρίνια θα μιλήσει. Είναι εκτελεστικός ε, διευθυντή ε, και εκπρόσωπος του Ισπανικού Δικτύου ε, με έδρα στην Μαδρίτη ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης θα σας διαβάσω το μήνυμα της ε, Μαδρίτης από τις γυναίκες με τα άσπρα. Η κυρία Σολέρα ήθελε να έρθει για να συμμετάσχει στη σημερινή συζήτηση, αλλά δεν μπόρεσε να ταξιδέψει. Θα το διαβάσω το μήνυμά της. Χαιρετίζουμε τους φίλους μας ε, στις Βρυξέλλες που μας δίνουν φωνή. 74 ε, ε, Κυριακές τώρα μας έχουν περικυκλώσει οι κυβερνητικοί και παραστρατιωτικοί που μας συλλαμβάνουν, μας χτυπούν, μας κακοποιούν για να μας αφήσουν να πάμε στη λειτουργία της Σάντα Ρίτα. έχουν περικυκλώσει την εκκλησία και δεν μπορούμε να μπούμε. Θέλουμε να επικεντρωθείτε κι εσείς σε ε, κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Φυσικά, ε, καταγγέλουμε ε, το περιεχόμενο συμφωνίας που είναι για μας υποχώρηση. Θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής και να προβληματιστείτε. Για ποιον είναι η συμφωνία Αυτά τα επιχειρήματα που προβάλλετε συστηματικά για να δικαιολογήσετε τη συμφωνία, εμεί είμαστε οι Ευρωπαίοι, έτσι καταλαβαίνετε τι λέει. Αναποτελεσματικότητα τη κοινή θέση. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Η κυρία Μπέρτα Σολέρ μα μιλάει για την αναποτελεσματικότητα, διότι προώθησαν ε, τις σχέσεις με τις ε, κουβανικές αρχές ε, χωρίς να απαιτήσουν σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έγινε σεβαστό το σύμφωνο αυτό. Δεύτερον, εξωτερική παρέμβαση. Οι κουβανοί θα πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Δεν, καμία εξωτερική παρέμβαση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Και ε, Σμεζόμαστε αυτό το επιχείρημα, αλλά δεν μας έλαβαν υπόψη και οι θύνοντες των κρατών μελών καθώς και υψηλή εκπρόσωπος συναντιόντουσαν και πέραν φωτογραφίες με τον Ραούλ Κάστρο ενώ αγνοούν την κατάσταση της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών. Μας αγνοούσαν να μην υπάρχουν. Ε, ε, θέλουμε να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση, θέλουμε να έχει την ηθική νομιμοποίηση που δεν έχει. Τρίτον, ε, η Κούβα και οι σχέσεις με τις χώρες της περιοχής. Η συμφωνία πλαίσιο για τις χώρες της περιοχής επίσης εφαρμόστηκε στην Κούβα χωρίς να λάβουμε υπόψη ότι η, η δικτατορία στην Κούβα είναι μόνο απολυταρχικό καθεστώ στην περιοχή και γι' αυτό δεν μπορεί να έχει την ίδια μεταχείριση. Ε, η, η περάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, φυσικά είναι, θα πρέπει να αποτελείται αντικείμενο της συμφωνίας ε, και θα πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστή νομοθεσία. Θα ήθελα επίσης να παραθέσω άρθρα του συντάγματος, άρθρο 3, όλοι οι πολίτες ε, μπορούν, έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν με όλα τα μέσα, ακόμη και με ένοπλο αγώνα, όταν δεν υπάρχει άλλο μέσο για να ανατρέψουν την πολιτική και κοινωνικονομική τάξη ε, του, που προβλέπεται από το Σύνταγμα αυτό. Επίσης, ε, ε, ο σοσιαλισμός και το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της Επανάστασης προβλέπεται από τον Σύνταγμα. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να επιτύχει την τα, μόρφωση της χώρας και να μας οδηγήσει σε μια δίκαιη κοινωνία. Ποια είναι τα συμπεράσματά μας. Ε, δίνεται το πράσινο φως στην κουβανική κυβέρνηση. Φαίνεται ότι τα συμφέροντά σας είναι με αυτούς που κερδίζουν. Τρίτον, το ευρωπαϊκό σχέδιο, παρότι νομοποιείται επίσης, ακολουθεί διαφορετική ε, κατεύθυνση σε σχέση με το δικό μας ε, διάβημα. Επίσης, η διεθνή κοινότητα είχε υποστηρίξει την ε, ειρηνευτική διαδικασία στην ε, Κολομβία. Ο Ραούλ Κάστρο όμω ε, δεν διευκόλυνε τη συμφιλίωση ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και παρατηρούν όλοι απαθείς αυτήν την πολιτική αδράνεια και την ταπείνωση του λαού της Κούβας. Αυτό λοιπόν με τον τελευταίο χαιρετισμό είναι το μήνυμα της κυρίας Σολέρο. Ε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Αντώνο. Δεν θέλετε κύριε Αντώνο, μάλιστα. Ο κύριος Γκυγέρμο τότε, Φαρίνας, υποψήφιος για το βραβείο Ζαχάρη το 2010. 6-7 λεπτά εισαγωγή. Okay. Ε, Ευχαριστώ πολύ. κυρίε και κύριοι βουλευτέ τη Ευρωβουλή. Είναι τιμή και υποχρέωση για μένα ως βραβείο Σαχάροφ να είμαι εδώ μπροστά σα, για να σας μεταβάσω τις ανησυχίε μου σε σχέση με την διμερή σχέση Κούβας ΕΕ που θα πετυχαίνει το στόχο που όλοι θέλουμε δηλαδή τον εκδημοκρατισμό της Κούβας ως αποτέλεσμα της πρόσπισης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων ως βάση συνύπαρξης, πρόοδου και ελευθερίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε και συνεχίζει να αποτελεί αγγιητή αυτών των δικαιωμάτων και θα πρέπει να συνεχίζει να το πράττει αυτό πέρα από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Σε αυτό λοιπόν βασίζεται το κύρος που ο θεσμός, σας, ο θεσμός Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνει διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα κύριο παράγοντα, ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές σύγχυσης για την ιστορία της Κούβας, για το κοβανικό καθεστώς το οποίο χρειάζεται νομιμοποίηση και πόρους. Ιδιαίτερα τώρα λοιπόν που βλέπει να τελειώνει η χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα. Ενώ για τους δημοκράτες της Κούβας αυτό που προέχει είναι η πρόσπιση των αξιών που εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι θεωρούν ότι η αλλαγή στην Κούβα θα έρθει μέσω της οικονομικής οδού. Εμείς σεβόμαστε αυτούς που έχουν αυτή την άποψη. Παρ' όλα αυτά, η κοβανική οικονομία ελέγχεται από μια στρατιωτικό-οικογενειακή ελίτ, η οποία διαχειρίζεται ολόκληρο το οικονομικό και εμπορικό σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, οι υποτιθήμενες μεταρρυθμίσεις, ακόμα και στον οικονομικό τομέα, είναι πολύ πτωχές και δείχνουν την αυταρχική φύση του καθεστώτος επειδή εφαρμόζει ακριβώς μια επίθεση στους μικροεπιχειρηματίες. Μικροεπιχειρηματίες που αυτοί φημιστικά επωνομάζουν μικροϊδιοκτήτες. Έχουν αρνηθεί λοιπόν να λάβουν κονδύλια για την ενίσχυση των μικρών επιχειρηματιών. Και ενώ μιλάμε εμείς εδώ έχουμε ένα κύμα καταστολής και κλεισίματος πολλών επιχειρήσεων μικροεπιχειρηματιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσει την ανάπτυξη αυτών των μικροεπιχειρηματιών και όχι να στηρίζει το κουβανικό καθεστώς με την τωρινή νομοθεσία. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση η κυβέρνηση θα είναι ο αποκλειστικός κύριος της οικονομίας της Κούβας. Θα ήθελα να μιλήσω και για τους εργάτες στην Κούβα και τους εργαζόμενους, των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται συνεχώς και συστηματικά. Αυτό συμβαίνει και στην Πορτογαλία, όπου έχουμε ένα μικρό ποσοστό ως αμοιβή 3 με 7% των αμοιβών που έχουν συμφωνήσει οι δύο χώρες. Αυτό αποτελεί μια εκμετάλλευση στην εποχή μας. Πώς γίνεται λοιπόν εμείς που θέλουμε να προσπίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων να είμαστε διάφοροι και αδρανείς μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα η οποία ούτε καν αναφέρεται στην συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προσπαθήσει να κατανοήσει ότι οι ηθικοί και πολιτικοί κώδικες του συνομιλητή της, δηλαδή της κουβανικής κυβέρνησης, δεν είναι αξιόπιστοι. Και για άλλη μια φορά δεν τήρησαν τα συμπεφωνημένα. Παραγματος χάρη στις συμφωνίες με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Νομίζω είναι αντίφαση το ότι στο πρώτο, του άρθρο, στο πρώτο της άρθρο συμφωνία κηρύσσει ότι ακριβώς τα μέρη θα προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και στη συνέχεια, αμέσως μετά, νομιμοποιεί το, το, το, το τωρινό νομικό καθεστώς, νομικό πλαίσιο μάλλον, του κουβανικού καθεστώτος, το οποίο είναι από τα χειρότερα στα ελληνικά καθεστώτα που υπήρξαν ποτέ. Κατά διάρκεια της ε, επισκεψής μας μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι δεν υπήρξε διαβούλευση με τους ευρωβουλευτές κατά διάρκεια της διαπραγμάτευσης της συμφωνίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους της κουβανικής κυβέρνησης και ενημέρωσης εκ μέρους της ΑΕΔ νομίζω αφορά την αξιοπιστία όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, Κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων η κουβανική κυβέρνηση απείλησε ακτιβιστές στο Πιναδελδρίο και οι γυναίκες στα Λευκά συνεχίζουν κάθε Κυριακή να δέχονται επιθέσεις και σωματική βία. Ενώ είχαμε λοιπόν την, διαπραγμα... την διαπραγμάτευση της συμφωνίας, οι ακτιβιστές συνέχισαν να δέχονται σωματική βία στην Αβάνα. Ενώ λοιπόν συνεχιζόταν η διαπραγμάτευση, αντιφρονούντες στην Αβάνα δέχτηκαν επιθέσεις και δίμευσαν τα, τα περιουσιακά του στοιχεία. Επίσης χτύπησαν και άλλους αντιφρονούντες επειδή μοίραζαν τρόφιμα και ε, βοηθούσαν τους πιο φτωχούς στη Βία Κλάρα. Και ενώ γινόταν διαπραγμάτευση, άτομα από την ε, Πατρική Ένωση της ε, Κούβας δέχτηκαν επιθέσει και κόντεψαν να, να πεθάνουν από, από τη φωτιά στη, σε ένα μέρος, σε μια πόλη τη Κούβα. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια στάση μια κυβέρνηση η οποία είναι τελείως ληστρική, ε, συμπεριφέρονται σαν κακοποιοί. Εσείς είσαστε άνθρωποι αξιοπρεπείς που ενεργούν καλή την πίστη. Πάντως να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία στις κουβανικές αρχές θα περιλαμβάνει προθεσμίες και δεσμεύσεις οι οποίες δεν θα τηρηθούν. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω. Αυτές τις μέρες βλέπουμε να επανέρχεται ένα ερώτημα και το αντιμετωπίζω και εγώ στο μυαλό και στη συνείδησή μου, Τι θα έπρεπε να πω στους ευρωβουλευτές από τη στιγμή που εσείς δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τη συμφωνία αυτή. Σας παρακαλώ να την καταψηφίσετε. Να την καταψηφίσετε ώστε να επαναδιαπραγματευτεί μια νόμιμη συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να μην πέσουν στο κενό αυτές οι εκκλήσεις. Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η ελευθερία όπως αυτή ακριβώς που ζούμε στις χώρες της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία σας. Θα δώσω τώρα στο λόγο στον κύριο Αλεχάνδρο Κονσάλ Έχετε παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέλη της Υποπιτροπής, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δίνεται σήμερα στο, στο Κουβανικό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να σας μιλήσει και να συζητήσουμε ακριβώς την συμφωνία που θα καθορίσει τις μελλοντικέ σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Κούβας. Δεν έχουμε να κάνουμε με σύνθεση διαδικασίες και αυτό το αισθάνονται και εκατομμύρια κουβανοί γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τις σχέσεις Κουβάς Αυτό που θα συζητήσετε σε λίγες ημέρες είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει στον κουβανικό λαό το δικαίωμά του να προασπίσει και να απολαμβάνει τον ίδιο δικαιωμάτων που απολαμβάνετε εσείς. Ή αντίθετα, αν θα συμβάλλουμε στην υποστήριξη μιας δικτατορίας που σύντομα θα συμπληρώσει 59 χρόνια αυταρχικού ελέγχου. Σύντομα λοιπόν θα αποφασίσετε αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια βία ηθικής στην Κούβα ή αν θα πρέπει να πράξουμε διαφορετικά. Έχουμε την έκθεση Μπίκερ Πακ ή και το μνημόνιο Σαραπάτ τη δεκαετία του 70 και αργότερα με τα κριτήρια της ε, Κοπεχάγης τη δεκαετία του 90. Επιτρέψτε μου να σας επιθυμίσω κάποια σημεία που περιλαμβάνουν αυτά τα έγγραφα. Η έκθεση λοιπόν Μπίκελπακ για τις ε, πολιτικές και θεσμικές ε, πτυχές έλεγε ότι καμία χώρα δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτή αν δεν είναι δημοκρατική στην κοινότητα. Και λέει το μνημόνιο Σαραγκάτ ότι η προσχώρηση αποκλείεται για τις χώρες των οποίων το πολίτευμα διαφέρει ουσιοδός με το πολίτευμα των υπολείπων χωρών. Αυτό βοήθησε αργότερα τις χώρες όπως η Ισπανία να προχωρήσουν στο δρόμο του εκδημοκρατισμού και να προσχωρήσουν στην Ένωση. Επίσης πρέπει να πούμε ότι είχαμε και τα κριτήρια της Κοπεχάγης που εγκρίθηκαν το 1993 για να επιτρέψουν τη μετάβαση των νέων υποψηφίων της Ανατολής προς την δημοκρατία. Εκεί καθοριζόταν επίσης και η πρόβλεψη για σταθερές δημοκρατικές αρχές που θα ασφαλίζει την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό των μειονοτήτων. Είναι προφανές ότι η, Κουβανία, η, συγγνώμη, η Κούβα επουδενή δεν μπορεί να αποτελεί υποψήφιο σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια. Βεβαίω θα πρέπει να συνεχίζουμε τι προσπαθίε μα για τον εκδημοκρατισμό τη. Ποτέ δεν θεωρήσε η Ευρώπη ότι για να έχει επιρροή σε αυτές τις χώρες θα έπρεπε να απαιτήσει συγκεκριμένα βήματα προς τον εκδημοκρασμό. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Οπότε το ερώτημα παραμένει, ξαναλέω, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να απολέσει την δημοκρατική της δέσμευση και την ηθική της δέσμευση προς τον κουβανικό λαό με αυτή τη συμφωνία. Γιατί θα κάνουμε διαφορετικά πράγματα από ό,τι κάναμε με άλλες χώρες επιτυχώς Κυρίε και κύριοι, αν θέλετε να γνωρίσετε την ε, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σα κάποια πράγματα. Η επανέναξη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΙΠΑ και Κούβα ήταν το αποτέλεσμα ενό αγώνα όπου κερδίζει αυτό που κάνει περισσότερε παραχωρήσει το καθεστώ. Αλλά στο τέλο κερδίζει πάντοτε το καθεστώ. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά είχαμε βέβαια και την επιβράβευση παγκοσμίω δημοκρατικών θεσμών όπως Ευρωπαϊκή Ένωση, ΙΠΑ κλπ. Είχε βέβαια και την έγκριση του Βατικανού αυτή η συμφωνία. Στην Κούβα όμως το πλαίσιο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μικρών δικαιωμάτων ενισχύεται ε, ενώ αυξάνεται η απόγνωση στη χώρα μας, η, κατα... η κατάφορη παραβίαση δικαιωμάτων έκφρασης, ε, συναθρίζεστε κτλ. Υπάρχει στο ίδιο το σύνταγμα τη Δημοκρατίας που λέει στο άρθρο 5 ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας μαξιστικό, λενινιστικό αποτελεί την διευθύνουσα δύναμη του κράτους η οποία διαργανώνει την κοινή προσπάθεια του λαού για την επίτευξη του σοσιαλισμού και την πρόοδο προς την κομμουνιστική κοινωνία. Αυτό το άρθρο, αυτό το άρθρο αρνείται τη συμμετοχή στα κοινά πράγματα αυτών που δεν επιθυμούμε τον κομμουνισμό ως πολιτικό σύστημα. Σε ένα άλλο άρθρο διαβάζουμε ότι αναγνωρίζεται στους πολίτες το δικαίωμα έκφρασης σύμφωνα με τους στόχους της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Δηλαδή, εκτός αυτού πλαισίου δεν υπάρχει δυνατότητα έκφρασης, ελεύθερης έκφρασης. Διαφορετικά, διαθέτει κανείς τον κύριο να φυλακιστεί λόγω έκφρασης. και αυτά εφαρμόζονται. Από το Δεκέμβρη είχαμε 16.000 παρόνομες συλλήψεις με αντίστοιχες παραβιάσεις ατομικών ελευθεριών. Δεκάδες κουβανοί εγκατέλειψαν τη χώρα από τα δάση ή από τη θάλασσα αναζητώντας την ελπίδα. Πολλοί όμως, πολλοί όμως βρήκαν το θάνατο. αρνούνται σε ανήλικους και σε γυναίκες να συμμετάσχουν σε δημοκρατικές πράξεις. Συνεχίζουν να χτυπούν άντρες και γυναίκες αδιάκριτα. Συνεχίζουν να παρεμβαίνουν στα κέντρα εργασίας, στην δουλειά τους ή προσπαθούν να καταστήλουν εναλλακτικέ οργανώσεις, επεμβαίνουν στα μέσα επικοινωνίας στιγματίζοντας την ελεύθερη έκφραση και την ελεύθερη σκέψη. Έχουμε δημεύσεις περιουσιών και το ανέφερε προηγουμένως ο Γκυλιέρμο είχαμε την Λαρίσα Ριβερσέν, την ε, δικηγόρο από μια ένωση που παρέχει δωρεάν δικηγορικές υπηρεσίες στο, στο λαό τις αρνήθηκαν την ε, είσοδο στη χώρα και αυτό αφορούσε και την οικογένειά της. Ο διάλογος πρέπει να αποτελεί το, τη μόνη λύση για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση. Βλέπουμε όμως ότι ο διάλογος δυστυχώς μεταμορφώνεται σε έναν βολονταρισμό ο οποίος καλύπτει και επιβάλλεται στις καλές προθέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε πολλές καλές προθέσεις και γενικές παγκόσμιες αρχές δύσκολα θα μπορούσε κάποιος δημοκράτης να διαφωνήσει όμως σε συγκεκριμένα ζητήματα, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Πάντοτε βλέπουμε ότι κάθε χώρα είναι ελεύθερη στην επιλογή του πολιτικού της συστήματος, το οποίο στην πράξη μεταφράζεται σε νομιμοποίηση της κυβουβανικής κυβέρνηση στην ε, καταστολή και στην έλλειψη ελευθεριών. Είναι ένα έγκλημα το να προσπαθήσει κανεί να νομιμοποιήσει αυτή την κατάσταση, λέγοντα ότι εμεί οι Κουβανοί ελεύθερα επιλέξαμε αυτό το σύστημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι κανένας στον κόσμο εθελοντικά, μάλλον θα μπορούσε από μόνος να επιλέξει την απώλεια, τη μη ύπαρξη ελευθερίας. Μετά από δεκαετίες επαφών και συνομιλιών με την Αβάνα βλέπουμε να αντιλαμβάνονται εκεί τα δημοκρατικά δικαιώματα με διαφορετικό τρόπο. Η συμφωνία λοιπόν αυτή δεν είναι η συμφωνία που χρειαζόμαστε. Λείπουν εγγυήσει, λείπουν μηχανισμοί συγκεκριμένοι που θα επιβάλλουν στην κουβανική κυβέρνηση την εφαρμογή αυτών των αρχών. Θα μας πούν βέβαια αυτοί ότι οι μηχανισμοί θα πρέπει να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν. Όμως ξέρουμε ότι αν από την αρχή δεν υπάρχουν οι απαραίτητε προβλέψει και εγγυήσει, τα πράγματα θα πάνε στη λάθο κατεύθυνση. Έχουμε κάποιες προτάσεις που θεωρούμε θα πρέπει να ενταχθούν στην συμφωνία αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τον πανικό λαό. Αυτές είναι κάποιες από τις ε, σκέψεις μας. Καταρχάς ότι θα πρέπει να αποκλείονται κυρώσεις ποινικέ ή διοικητικές που θα τιμωρούν τους πολίτες ε, στην άσκηση των ε, πολιτικών του δικαιωμάτων. Οπότε θα πρέπει να απαιτηθεί η άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και η πάυση τη αστυνομική βία. Η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή όλων των διεθνών συμφωνιών όσον αφορά τα δικαιώματα, τα ατομικά και τα συλλογικά. Η συμφωνία επίση θα πρέπει να καθορίζει διαλόγου, συνομηχανισμού, πολιτικού πολιτικού διαλόγου με την ανεξάρτητη και ελεύθερη κοινωνία των πολιτών στην Κούβα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός ώστε όλοι οι πολίτες να είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να είναι σε θέση να καταγγέλουν, να καταγγέλουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αρχών. Θα πρέπει επίση να αποκλείσουμε οποιαδήποτε μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης μια πρακτική η οποία είναι συστηματική από το κουβανικό κράτος ιδιαίτερα όσον αφορά το πλαίσιο των ξένων επενδύσεων. Επίσης, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στην ε, Κούβα θα πρέπει να εφαρμόζουν τις ίδιες αρχές που εφαρμόζουν στις χώρες τους, ιδιαίτερα αυτές που λαμβάνουν κονδύλια ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομική βοήθεια δημόσιας φύσης. Η συμφωνία επίσης θα πρέπει να ζητά την πάυση τη διακριτική ευχέρεια τη κουβανική κυβέρνηση για την είσοδο ή έξοδο των ίδιων των κουβανών πολιτών. Όσον αφορά τη διαδικασία τώρα τη συμφωνία, θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια μεταβατική διάταξη η οποία θα προβλέπει μια κλιμακωτή εφαρμογή στα διάφορα, στο διάφορα πεδία συνεργασίας που θα ακολουθεί την προπόθεση τη εφαρμογή αυτών των αρχών από την κουβανική κυβέρνηση. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια ρήτρα δημοκρατία, η οποία θα καθορίζει δικασίε και του τρόπου με του οποίου θα καταγγέλλεται αυτή η συμφωνία όταν θα υπάρχει συστηματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρίε και κύριοι, οι δημοκράτε τη Κούβα εργαζόμαστε για να πετύχουμε μια δημοκρατική κοινωνία με ευκαιρίε για όλου και μάλιστα χωρί να αποκλείσουμε αυτού που βρίσκονται στην κουβανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Είναι όμω απαραίτητο να μην υποχωρήσουμε στι απαιτήσει μα, στι διεκδικήσει μα, ώστε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ελευθερία να είναι σεβαστέ. Η Κούβα δεν ανήκει μόνο την κυβερνητική ελίτ όσο και αν προσπάθησαν πάνω από μισό αιώνα να το πετύχουν αυτό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει αυτές οι απαιτήσει, αυτές οι περιποθέσεις να καταγραφούν στη συμφωνία και να ζητήσουμε σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχή διάλογο με τους κουβανούς και μεταξύ των κουβανών. Κυρίε και κύριοι, έχετε μπροστά σας το μεγάλο δίλημα. Να αναγνωρίσουμε αυτά τα δικαιώματα ή να καθορίσουμε ένα είδο απόρριψη βασικών αρχών εκ μέρου αυτού του σώματο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα οι συναδελφοί. Η κυρία Αντρίκη για το ΕΛΚ. Λάιμα, ΕΛΚ. Εσύ είσαι στο ΕΛΚ, το, το κόμμα σου είναι. Θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου που βλέπω τον Κόκο στο Ευρωκοινοβούλιο και πάλι. Πριν μερικά λεπτά ακούσαμε δύο πολύ ισχυρές δηλώσεις. Μία από τις κυρίες Μεταλλευκά και μία από τον υπόλοιπο υποψήφιο για το Σακχάροφ τον Φαρίνια. Δύο βασικές δηλώσεις που απευθύνονται στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης που κάνουν λόγο για την εξοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο και που έχει σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας. Έχω δύο ερωτήματα να θέσω στον Κιέρμα Φαρίνιας όπως όλοι γνωρίζουμε, το άρθρο 2 σε όποια συμφωνία εταιρική σχέση ε, και συμφωνίας αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αν οι διαπραγματεύσει ε, συμπεριλαμβάνουν και δημόσιες διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, θα ήθελα να είμαι βέβαιη να μας δώσετε πληροφορίες αν όντως λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους διαβουλεύσεις στην Κούβα. Το δεύτερο ερώτημα είναι... Ε, αφορά την ε, αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αβάνα. Λάβατε πρόσκληση για να συναντήσετε τον επικεφαλής της αντιπροσωπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ξεκίνησε τι εργασίε τη υπηρεσβείας στην ε, Αβάνα. Λάβατε πρόταση. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Σασής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχίζοντας να χαιρετήσω τους κυρίους ε, Φαρίνιας ε, και Κονσάλης Ράνια και κυρίως τον κύριο Φαρίνιας. Στη Λισαβόνα συναντηθήκαμε πριν από λίγους μήνες και τότε ε, εξέφρασε τη λύπη του διότι η πορτογαλική κυβέρνηση ε, ούτε και η δική του κυβέρνηση μπόρεσαν να εκφράσουν ε, τη βούλησή τους για να λάβει το βραβείο Ζαχάροφ. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για την προσπάθεια που έχετε κάνει. Έχετε κάνει επανειλημμένα απεργία πείνας, έχετε θέσει εν κινδύνο τη ζωή σας για να υπερασπιστείτε τις αξίες που είναι και οι θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και πιο συγκεκριμένα η ελευθερία. Κάποιοι ε, κάνουν ότι το αγνοούν, αλλά εσείς όχι. Εξακολουθεί να είναι μαρξιστικό, λενινιστικό, απολυταρχικό καθεστώς αυτό της Κούβας. Και είναι και το τελευταίο που υπάρχει στον κόσμο. Με αυτό το άνοιγμα από πλευρά των ΗΠΑ και το άνοιγμα από πλευρά της Ευρώπης μπορεί να επέλθει και μια αλλαγή της κοινωνίας. Ε, όπως είπε και ένας αλφούς ε, πριν από λίγα χρόνια, αυτό δεν είναι σίγουρο, ε, λίγες, ε, λίγα λεπτά, δεν είναι σίγουρο αυτό ότι θα συμβεί αυτό αυτό το οικονομικό άνοιγμα μπορεί να συνεπαθεί ένα, ένα εκδημοκρατισμό, όμως αν κοιτάξουμε στην Ισταρία μπορούμε να δούμε άλλα παραδείγματα όπου δεν επήλθε και πολιτική αλλαγή μετά από την οικονομική αλλαγή. Όσοι ζουν στην Κούβα, όσοι έχουν πέσει θύματα αυτού του ε, κατασταλτικού καθεστώτος, έχουν προσδοκίες σε σχέση με αυτές τις αλλαγές που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και ελπίζουν ότι ε, θα οδηγήσουν σε κοινωνικές αλλαγές και σε εκδημοκρατισμό. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ο δημοκρατισμός δεν πρόκειται να υλοποιηθεί αν εμείς οι ευρωβουλευτές δεν συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ε, τον αγώνα των κουβανών που ε, αγωνίζονται για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι απαραίτητο με πεποίθηση να ε, υποστηρίξουμε ε, αυτό που πιστεύουν οι βουλευτές, να σταθούμε στο πλάι σας σε αυτόν τον αγώνα. Και θα κλείσω εδώ λέγοντας ε, ότι μετά από αυτά τα ανοίγματα, μετά από την αλλαγή της αμερικανικής θέσης, μετά από τις προσδοκίες που υπάρχουν για αλλαγή, μπορείτε να μας πείτε εάν υπήρξε κάποια αλλαγή από πλευρά κουβανική κυβέρνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το διάλογο με αυτού που αγωνίστηκαν για να επικρατήσει ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπω εσεί, σα ευχαριστούμε, λέει ο κύριο Περέντα. Κύριε Μπεσέρα, για του φιλελεύθερους. Ε, Αλεχάνδρο, καλώς ήρθες ε, και πάλι. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμά σου. Θέλω να θυμίσω και πάλι ότι αυτή η συμφωνία με την Κούβα είναι η πρώτη διμερής συμφωνία και αυτό δείχνει ένα ε, ρεαλισμό ε, που χαρακτηρίζει την πολιτική και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κόσμο. Για θέματα ασφαλείας αυτός ο ρεαλισμός συμμορφώνεται, συνάδει με αυτήν τη νέα θέση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να σταματήσουν οι κενές υποσχέσεις όπως με αυτό το σύμφωνο. Θέλουμε στην πράξη να εφαρμοστούν ε, αυτά που έχουν αποφασιστεί. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα σημειωθεί η πρόοδος, θα γίνουν βήματα και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην συμφωνία θα πρέπει να αναφερθούν αυτά και είναι ε, σημαντικό να αναφέρονται και να περιέχονται στη συμφωνία. Ακόμα σημαντικότερο όμως είναι να εφαρμοστούν. Μιλάμε για εθνικούς μηχανισμούς ε, και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να του επηρεάσουμε τους ώστε να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή σε σχέση με αυτά που μας είπες και εσύ τώρα. Πιστεύεις ε, πως η αξία του βραβείου Ζαχάροφ που απενέμεται στο Κοινοβούλιο, γιατί για μας είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πιστεύεις ότι ενισχύεται η αξία του βραβείου Ζαχάροφ και υπάρχουν τρία, σε τρία βραβεία Ζαχάροφ ε, στην Κούβα. Πιστεύεις ότι αυτό έχει κάποια σχέση με τις προσδοκίες? Ότι δηλαδή σας δίνει μια φωνή το Κοινοβούλιο και ε, εστιάζουμε στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με αυτά τα ε, τρία βραβεία Ζαχάροφ που έχουν απονεμηθεί τα τελευταία 28 χρόνια πιστεύεις ότι ε, έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πόρους ε, στην ε, Κούβα και πιστεύεις ότι δίνεται μια φωνή σε αυτούς τους ανθρώπους ή πρέπει να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία. Πρέντα, ε, άλλοι δύο, τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που κάνετε την προσπάθεια. Υπάρχουν δύο σχολές στο να δούμε την συμφωνία. Η μία σχολή ότι αυτή η συμφωνία θα πρέπει να οδηγήσει σταδιακά σε αλλαγέ στη Γη. δεύτερη σχολή είναι, έχει αμφιβολίε. Δεν σα πω ποια είναι σωστή από τι δύο, αλλά όταν διάβασα για πρώτη φορά το σχέδιο τη συμφωνία, χωρί να έχω υπερβολικέ προσδοκίε, πρέπει να πω ότι σοκαρίστηκα. Ήμουν μέλο τη αντιπροσωπεία για τι πρώτα στα διαπραγματεύσεων, την πρώτη ε, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Τσεχοσλοβακίας και μετά συμμετείχα στις ε, συζητήσεις ε, για την προσχώρηση. Μετά το 1989, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επισκεφθεί την Κούβα αυτό που με εντυπωσιάζει και πιστεύω ότι θα βρεθεί μια ισορροπία σε αυτό, δεν υπάρχει μία, μια παραμικρή δέσμευση για την Κούβα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ούτε μία δέσμευση. Όλες οι διατάξεις έχουν ε, συνταχθεί με αναφορά σε διμερείς σχέσεις και ότι θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για εμένα αυτό είναι είναι υπερβολικά απογοητευτικό. Και μια άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω για να τονίσω τι είδους διάλογο για τη κούβα να έχει μα, εμάς. Τον αντιπρόεδρο ε, του Άλμπε θέλω να ρωτήσω για τις συζητήσεις που είχε στην Κούβα. Ο συνάδελφος Ζωζέ ήταν ένα άλλο μέλο, μέλος πολλές φορές μας ε, διατυπώθηκε ότι δεν είμαστε ευπρόσδεκτοι γιατί τα τελευταία χρόνια και πριν 10 χρόνια που μπήκαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφραστήκαμε και εγκαταστηθήκαμε ως προς τα στην παραβίαση των δικαιωμάτων στην Κούβα. Τέτοιου είδου πολιτικό διάλογο έχουμε σήμερα, όπω καταλαβαίνετε. Και το τρίτο θέμα που θέλω να θίξω έχει σχέση με, μια συνέντευξη που είχαμε με δύο άλλους ε, συναδέλφους με αξιωματούχους ε, της επιστημονικής δράσης συν τον πρέσβη όπου μας είπαν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην Κούβα ότι είναι υπερασπιστές ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό όμως είναι κάτι που ίσως εσείς, όχι μόνο εσείς, και άλλοι συναδελφοί σας άλλους ε, συνδυασμούς, γιατί συναντούμε διάφορους αντιφρονούντες κτλ. Μέσα από την οπτική κάποιου που είναι υπέρ της αντιπολίτευσης, δεν βλέπουμε την ενότητα που θα θέλαμε να έχουμε από την πλευρά σας, όχι ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ως ηγέτες της αντιπολίτευσης και να αναπτύξετε τον διάλογο, ότι δεν έχει αναπτύξει τον διάλογο με τις αρχές, αυτών που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ για τη σύντομη παρέμβαση, κύριε Φαριά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα τα πω πρωτοκαλικά. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Φαρίνιο ε, και ε, το κύριο Κονσάλες ε, και την κυρία Λανινάγκο που ήρθανε σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, ευχαριστώ για το κουράγιο που δείχνετε. Έρχεστε εδώ πέρα για να καταγγείλετε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή ε, στην Κούβα, θέτοντας εν κινδύνο τη ζωή σας. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν θέλω να μιλήσω για το καθεστώς, ε, διότι ε, τα ακούσαμε από τους συναδέλφους. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που ακούσαμε. Θέλω να επαναλάβω κάτι που έχω πει και σε άλλες ε, συνεδριάσεις, ε, το λέω πάντα το δημόσιο, ότι αυτή η συμφωνία είναι επονίδιστη. Είναι μία συμφωνία που δεν λαμβάνει υπόψη διαστάσεις ε, που θα έπρεπε. Ανθρώπινα δικαιώματα, Φερπίν, πολιτικούς κρατούμενους, η πρέσβυρα δεν είναι εδώ, κρίμα, ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν ε, κρατούμενοι, υπάρχουν ε, ε, τρο, τρομοκράτες, μας λένε, αλλά πολιτικοί κρατούμενοι δεν υπάρχουν. Από τις αρχές του χρόνου, περίπου 8.000 άνθρωποι κρατήθηκαν. Ε, πρόκειται για, ε, μας λένε, εγκληματίες κοινού δικαίου, δεν είναι πολιτική κρατούμενοι, μας διαβεβαιώνουν. Χρειάζεται διαφάνεια, όπως είπε ο κ. Φαρίνιας. Και τελειώνω, τελειώνω, Πρόεδρε. Απλώς είναι σημαντικό να πω και ήδη το έχω ζητήσει με τον Υπουργό Υγεία μας στην Πορτογαλία. Είναι αυτό το ζήτημα των εργαζομένων, όπως είπε και ο κύριος Φαρίνιας. Αυτοί οι γιατροί, που, οι κουβανοί που ε, τους εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση. Αυτοί δουλεύουν στην Πορτογαλία. Και είπαμε τις 8.000 μεταναστών που, έχουν, που είναι εγκλωβισμένοι ανάμεσα στην Νικαράγουα και στην Κώστα Δεν αναφέρεται τίποτα μέσα στη συμφωνία. Έχουν φτιάξει ένα ε, ροζ χάρτη όπου δεν φαίνεται, της κατάστασης όπου δεν φαίνεται τίποτα από όλα αυτά. Κύριε Κονσάλες Ράγα, Κύριε Φαρίνιας, κλείνοντας να σας ρωτήσω, όπως είπε και ο συνάδελφος Φρανσίσκο Ασής, ε, πρέπει να έχετε την πεποίθηση ότι θα είμαστε σε εγρήγορση. Θα παρακολουθήσουμε από κοντά όλα αυτά που συμβαίνουν. Και ε, τώρα, Πρόεδρε, πραγματικά θα κλείσω. Ε, ο Σίκο Γκουαρκέ δεν ξέρω αν τον ξέρετε, ένας ε, ε, βραζιλιάνος ε, τραγουδιστής ο οποίος είπε για την Κούβα ότι θα γίνει μια μεγάλη Βραζιλία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι οι επαφές με στην καλή κατεύθυνση, σωστή κατεύθυνση. Κάποιοι λέγανε ότι κάποια θέματα δεν μπορούν να συζητηθούν και όμως ίσχυσε το αντίθετο. Είχαμε μια κοινή θέση της Ένωσης, στην οποία ηγήθηκε ο κ. Αθνάρ, ο πρώην Πρωθυπουργό, επειδή ήταν ανήκουστη. Νομίζω ότι μάλιστα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια ενδιαφέρουσα συμφωνία, σεβόμενη την κυριαρχία και των δύο μερών. Νομίζω ότι Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αποφάσεις των ΗΠΑ που αφορούν ευρωπαϊκές ε, τράπεζες, 8 δις ας πούμε πρόστιμο στην BMP κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν θα πρέπει να χειραγωγηθεί παρόλα αυτά από συγκεκριμένα άτομα, το οποίο όμως πραγματικά στην ουσία δεν ξέρουμε ποιον εκπροσωπούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και Πρόεδρος. Ένα λεπτάκι. Τέρεσα, Τέρεσα Χιμένες. Τελευταίος ομιλητής, έτσι. Θα προσπαθήσω να τα πω γρήγορα. Μίλησαμε τους προσκεκλημένους μας από χθε, αλλά να τους ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία τους. Ξέρω ότι ο κ. Φαρίνια ρισκάσει την υγεία του για την ελευθερία στην Κούβα ή και άλλοι φυλακίστηκαν σε φυλακές που δεν έχουν καμιά σχέση με αυτές τις φυλακές που έχουμε στην Ευρώπη. Να ευχαριστήσω και την Μπέρτα και όλες τις γυναίκες στα Λευκά που γνωρίζω επειδή ήρθαν να μας επισκεφτούν. Εσείς έχετε περισσότερη αξιοπρέπεια από όσοι θα μπορούσα να έχω εγώ όλη μου τη ζωή. Ξέρω ότι δεν είστε κατά μια ε, συμφωνία. Αυτό θα πρέπει να το επαναλάβουμε. Δεν είστε κατά μιας συμφωνίας Ένωση Κούβα. Δεν θέλετε όμως μια συμφωνία που δεν οδηγεί σε πραγματικά ανοίγματα. Σε μια συμφωνία η οποία δεν περιέχει συμβασμούς Ξέρω ότι άτομα όπως εσείς οι γυναίκες ε, στα Λευκά κατηγορήθηκαν για την αποτροπή συμφωνία με την Ένωση. Με την Ένωση. Δεν ισχύει όμως αυτό. Εσείς θέλετε να μην νομιμοποιηθεί μια αυταρχική κυβέρνηση, κάτι τελείω διαφορετικό. Αυτό που θα πρέπει να ρωτήσουμε ειλικρινά είναι ποιον ωφελεί αυτή η συμφωνία. Αν η απάντηση είναι τους κουβανούς, τότε εντάξει να το υποστηρίξουμε. Αν όμως αυτό δεν ισχύει, θα πρέπει να κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση όσον αφορά τη δέσμευσή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Τερέσα. Θα δώσω τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους μας, ο Αλχάνδρου Γκοσάλες πρώτα και μετά. Δεν ξέρω αν η ΕΔ θέλει να λάβει το λόγο και η ΕΔ. Ωραία. Ναι, Πρόεδρε. Η ΑΕΔ πρώτα. Και θα μπορούσε να μιλήσει, ο οποίος συμμετείχε άμεσα στις διαπραγματεύσεις. Αλλά πριν να του δώσω το λόγο, αν θέλετε, να σας πω ότι άκουσα με προσοχή όλες τις παρεμβάσεις. Και η διαδικασία αυτή δεν είναι σημερινή, αλλά ισχύει εδώ και χρόνια. Τους άκουσα όλους, κάναμε εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και θεωρούμε ότι η συμφωνία που έχουμε μπροστά μας είναι ισορροπημένη, επικοδομητική, αυστηρή, που περιέχει όλες τις προβλεπόμενες ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα πλαίσιο βελτίωσης των συμφερόντων και της Ευρώπης αλλά και της Κούβας. Και αν θέλετε θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο. Θα είμαι σύντομο. Θέλω απλώ να επανέλθω σε κάτι που ήδη έχει υποθεί στην αρχή. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ποιε είναι οι εναλλακτικέ. Να δούμε ποιε είναι οι εναλλακτικέ για την συμφωνία αυτή και να δούμε την κατάσταση τα τελευταία 60 χρόνια. Η Κούβα ήταν σε απομόνωση, απομονωμένη από τι ΗΠΑ κατά πρώτον, αλλά και ε, αποστασιοποιημένη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια. Και αυτή η πολιτική δεν βοήθησε να προωθηθεί το συμφέρον μας, τα συμφέροντά μας στην Κίνα. και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στην Κούβα. Γι' αυτό είναι καιρό τώρα να αλλάξουμε αυτή τη σχέση και να βρούμε άλλου επικοδομητικού τρόπου για να πετύχουμε του κοινού στόχου. Πρέπει να έχουμε μια καλύτερη πλατφόρμα, ένα καλύτερο πλαίσιο στο οποίο θα υπερασπιστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Η συμφωνία ορίζει τους όρους, τους τρόπους ε, με τους οποίους θα συνεργαστούμε με την Κούβα και θεωρούμε ότι αυτός είναι ο τρόπος για να πετύχουμε τους πολιτικούς στόχους στη σχέση μας με την Κούβα και από τη στιγμή που το PDCA είναι ένα εργαλείο για να επιδιώξουμε αυτούς τους στόχους, δεν θα ήταν σοφό να το υποβάλουμε σε όρους που θα μας στερήσουν την ύπαρξη αυτού του εργαλείου του μέσου. Μια άλλη ερώτηση που έχω να κάνω αφορά το άρθρο Ενα πέντε. Θα ήθελα να το κοιτάξετε. Η αναγνώριση του κουβανικού συντάγματος δεν είναι ακριβώς αυτό που ε, θα πρέπει να το διαβάσουμε προσεκτικά. Θα πρέπει οι δράσεις να ληφθούν σύμφωνα με το υπάρχον σύνταγμα, τις νομικές διατάξεις και με, σύμφωνα με τις συμφωνίες ε, σε διεθνές επίπεδο. Αυτό, επομένως, διέπει τη συμφωνία αυτή και η τελευταία παρατήρηση όσον αφορά την διαδικασία διαβουλεύσεων που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Προφανώς συμφωνούμε ότι η κοινωνία και τα μέσα μας θα πρέπει να ενημερωθούν για τις εξελίξεις που ε, υπάρχουν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κούβας και των τρίτων μερών. Αυτές οι διαπραγματεύσει γίνονται μεταξύ κυβερνήσεων και εκπροσώπων κυβερνήσεων. Θα πρέπει να ενημερώνονται λοιπόν και η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωση μέσω δελτίων τύπου και οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν συστηματική επαφή, επαφές ε, με τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες όσο και στην Κούβα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες και πολλές προσδοκίες από πολλούς τομείς της ε, κοινωνίας της Κούβας και αυτό φυσικά θα πρέπει να επηρεάσει τον ε, κύκλο των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Να πω έχουμε, να πω ότι έχουμε ότι είχαμε προσκαλέσει για την πρέσβυρα της Κούβας, αλλά είπε δεν μπορεί να έρθει. άλλες Ράκα τώρα. Και μετά θα κλείσουμε. Έχετε το λόγο. Να σας πω, απαντώντας σε αυτό που αναφέραμε εδώ, για την αξία των βραβείων. Θα μιλήσει καλύτερα ο Γιλιάρμο. Η πολιτική κρατούμενη είπε η πρέσβυρα ότι δεν υπάρχουν. Θα σας μιλήσω για ένα που γνώρισα στη φυλακή και παραμένει στη φυλακή. Επειδή χθε έλαβα ένα μήνυμα από το Αρμάντο Σόσα Φορτούνη έναν ε, κρατούμενο 73 ετών. Θα κλείσει 22 χρόνια στη φυλακή και είχε ήδη καταδικαστεί 14 χρόνια στη φυλακή. Είναι αλήθεια ότι μπήκε στην Κούβα μια νόπλη ομάδα που προσπάθησε να ανατρέψει την πολιτική τάξη στην ε, Κούβα. Όπως ακριβώς έκανε και η κουβανική κυβέρνηση, έτσι, με τον ίδιο τρόπο με ενόπλο τρόπο. Κατέλαβα την εξουσία. 22 συν 14 λοιπόν, ίσως να είναι ο πολιτικός κατούμενος που έχει πέρασει τα περισσότερα χρόνια στη φυλακή. Δεν αναφέρεται αυτό το περιστατικό συχνά γιατί δεν είναι πολιτικά correct. Αλλά έχουμε και τον Μπέρτο Ρέα που είχε καταδικαστεί σε θάνατο επειδή ακριβώς είχε λάβει μέρος στην ίδια διήστηση με την ίδια ενόπλη ομάδα που μπήκε στη χώρα καταδικάστηκε σε θάνατο κρατήθηκε 16 χρόνια αναμένοντας από μέρα σε μέρα την εκτέλεσή του μετάτρεψαν την ποινή του σε ισόβια τώρα Θα ρωτήσω λοιπόν η κουβανική κυβέρνηση που τόσα χρόνια καταπιέζει τους κουβανούς μήπως θα πρέπει να μας πει και αυτή την άποψή της. Εμείς είμαστε υπέρ της συμφωνίας πάντως. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία με την Κούβα. και θα στηρίξουμε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει αρχές που θα πρέπει να τηρήσει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει πραγματική βούληση προόδου στον πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η κουβανική κυβέρνηση. Αν αυτό ισχύει, γιατί φοβούνται. Γιατί δεν θέλουν να δεσμευτούν εδώ, σε αυτή τη συμφωνία. Αν και αυτοί επιθυμούν το ίδιο. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο εγώ. Bueno, ε, Ωραία. Να απαντήσω στην κυρία Λάιμα. Που και ευθυνής ο λαός υπέφερε από σταλινικό αυταρχικό καθεστώς. Να πω ότι εμείς δεν ρωτηθήκαμε ποτέ για αυτή, την τη συμφωνία και η οργάνωση που εκπροσωπώ η δεύτερη μεγαλύτερη και η πρώτη, με πιο πολύ αριθμή, η Πατρική Ένωση της Κούβας δεν ρωτήθηκε για την συμφωνία αυτή. Δεν υπήρξε ποτέ διαβούλευση. Μπορώ επίσης να σας μιλήσω εξ ονόματος των ε, γυναικών στα Λευκά, που είναι η πιο μεγάλη οργάνωση. Ούτε και αυτή ήταν ε, αντικείμενο διαβούλευσης. Ο κύριος Νάουτ είπε κάτι σχετικά και να πω εδώ ότι σε σχέση με το άλλο ερώτημα που είχαμε στις επαφές δηλαδή με την αντιπροσωπεία της Ένωσης στην Αβάνα τι να σας πω όσοι λάβαμε το βραβείο Ζαχάροφ δεν έχουμε μια προστασία από αυτό το βραβείο. Ίσως κάποια στιγμή να χρειαστεί να κρατήσετε ένα λεπτό σιγή για μένα. Είχαμε και άλλα άτομα τα οποία δέχτηκαν επιθέσει και είχαν λιποθυμίσει μετά από επιθέσει και είχαν πάρει το βραβείο Ζαχάροφ. Οπότε δεν υπάρχει καμία προστασία το βραβείο Ζαχάροφ του Κοινοβουλίου, να σα το τονίσω αυτό. Έχουμε στείλει τέσσερι επιστολέ στώντας από τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Ένωσης στην Αβάνα να μας ε, συναντήσει και δεν καταδέχτηκαν να μας απαντήσουν. Δεν πήραμε καμία απάντηση οι τέσσερις αυτές οργανώσεις, έτσι που στείλαμε επιστολές. Ο προηγούμενος επικεφαλής είχε επαφές, επαφές μαζί μας για να, δούμε, για να εξετάσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό γίνονταν τακτικά μετά από αιτήματά μα. Ο κύριο από την Πορτογαλία, ο ευρωβουλευτή, μας ρώτησε ο κύριο Ασή, τι γίνεται με το άνοιγμα με τι Ηνωμένες Πολιτείες, ποια είναι η κατάσταση, πώς συμπεριφέρεται η κυβέρνηση. Χειρότερα είναι η απάντηση. Υπάρχουν περισσότερες φυλακίσεις, περισσότερες απλές θανάτου, περισσότερες συλλήψεις. Ήδη έχουν τριπλασιαστεί κιόλας ή τετραπλασιαστεί. Και υπάρχουν περισσότεροι ύποπτοι. Θεωρεί λοιπόν το καθεστώς ότι νομιμοποιείται από τη ΣΥΠΑ και την Ένωση Μιλάμε για άτομα στην κυβέρνηση που έχουν νοοτροπία κακοποιών, μαφιόζων. Αυτός που έχει την εξουσία στην Κούβα σε μια επίθεση σε ένα στρατόπεδο σκότωσαν περισσότερα άτομα από ότι οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένο στην Κούβα αλλά ο τερνός ηγέτης της Κούβας έκανε επίθεση σε ένα νοσοκομείο θέτοντα σε κίνδυνο τη ζωή ασθενών, γιατρών, νοσοκόμων. Το νοσοκομείο αυτό, Σατουρνίνο, ήταν αντικείμενο επίθεση από τον Ραούλ Κάστρο, δηλαδή αυτά τα άτομα έχουν καμιά ακριβώς αντίσταση, καμία αμφιβολία να κάνουν οτιδήποτε για να πάρουν την εξουσία και να την κρατήσουν στα χέρια τους. Αυτό ως απάντηση προς τον κύριο Ασής. Για την κυρία Μπεθέρα να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι ουσιώδες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη έγινε ένα σημείο αναφοράς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω. Γιατί μετά το ολοκαύτωμα εσείς βρεθήκατε σε μια κατάσταση όπου χρειάστηκε να αποφασίσετε να θεσπίσετε κάποιους κανόνες ώστε τα ανθρώπινα όντα να μην σφάζονταν πια. Αυτό λοιπόν το σημείο αναφοράς ηθικής και το Κοινοβούλιο μέσω αυτού τρεις φορές απένιμε το βραβείο Ζαχάροφ. Αλλά θεωρούμε ότι μας εγκαταλείψατε όταν κάνουμε καταγγελίες καταγγελίες με κίνδυνο της ζωής μας και των οικογενειών μας. Δεν λαμβάνονται λοιπόν υπόψη αυτές οι καταγγελίες και υπερισχύουν οικονομικά συμφέροντα και ηγεμονικά συμφέροντα παραβλέποντας μια βασική αρχή ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα υπερέχουν των πάντων. Μπορούμε να πούμε στο φίλο εδώ που απουσιάζει ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα και αυτό είναι ένα θέμα σε κρεμότητα και σας καλώ να διαβάσετε την εφημερίδα Vanguardia από την περιφέρειά μου και θα δείτε ένας απόστρατος στρατηγός της ασφάλειας, της κρατικής ασφάλειας κομπάζει ότι είχαν δημιουργηθεί ομάδες θανάτου για την δολοφονία ακόμα και ανηλίκων με τη βοήθεια Ρώσων. Όπως και δηλαδή αυτοί στη χώρα τους ή και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως την Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία κλπ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Φαρίας για την ενθάρρυνση και την ελπίδα που μας προσφέρει. Θα προχωρήσουμε λοιπόν, έστω με κίνδυνο της ζωής μας, επειδή η ευημερία της πατρίδας δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με κανέναν. Για τον κύριο Κόουσο να πω ότι με κάθε σεβασμό να πω ότι ως δημοκράτες σεβαζόμαστε την άποψή του. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά ο πατέρας μου, να πω, ήταν μέλος του κινήματος 26 Ιουλίου. Και η μητέρα μου που είναι εδώ. Και ο Φιδέλ Κάστρο με μία απόφαση επέβαλε τα τρία μηδενικά. Μηδέν ε, μουσική, μηδέν ε, ε, κινηματογράφο, μηδέν θεάματα, για να μην υπάρχει ψυχογεία για το λαό. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι τρομοκρατία, τότε τι είναι τρομοκρατία. Αν εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι είναι επονίδιστο να έχουμε μια κοινή θέση, τότε ακριβώς θα πρέπει να δούμε το χαρακτηρισμό Γι' αυτό, για αυτή την κρατική τρομοκρατία εις βάρους του ίδιου του λαού που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Φιντέλ και του Ραούλ Κάστρο και του Αλεχάνδρο Κάστρο κιόλα, ο οποίος ε, είναι αυτός που έχει την πραγματική εξουσία αυτή τη στιγμή στην Κούβα. Στα 17 μου πήγα στην Αγκόλα και φέρω δύο τραύματα. Ήμουν μισθοφόρος υπέρ της Εσουσουδού. Και νομίζω ότι πολλοί από αυτούς τους στρατιώτες εξαφανίστηκαν. Αυτό νομίζω πολύ περισσότερο, πολύ πιο επονίδιστο από την κοινή θέση. Να ευχαριστήσω και την Τερέζα Χιμένες Να ευχαριστήσω λοιπόν Τέρεζα Χιμένες για την στήριξη, για την κατανόηση του αγώνα μας. Αυτές τις τρεις μέρες καταλάβαμε ότι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ακόμα πολλά σε επίπεδο αξιών. Θεός να σε ευλογεί και να ξέρετε ότι δεν θα μετανιώσετε ποτέ για το βραβείο που μου απονείματε, γιατί να ξέρετε ότι θα δώσω και την τελευταία πνοή της ζωής μου, ώστε στην Κούβα να έχουμε το ίδιο σύστημα, ώστε να μπορούμε να συζητάμε ανοιχτά και ελεύθερα με την ε, κυβέρνηση, με το ίδιο σύστημα δηλαδή που έχετε και εσείς στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας. Λυπάμαι για τους συναδέλφους που θα ασχοληθούν με το επόμενο θέμα γιατί έχουμε καθυστερήσει. Δεν ξέρω, θα μας πει ο κ. Φαρίνα, θα συνεχίσουμε τη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ. Señores, vamos a Θα συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο. Παρακαλώ. Καθίστε. Δεν με ακούει κανείς, λέει η Πρόεδρος. Θα ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα. No eh, Παρακαλώ κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ξεκινήσουμε. Για άλλη μια φορά. Θα συζητήσουμε την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Απόδειξη του μεγάλου ενδιαφέροντος του σώματος για το λαό της Βενεζουέλας. μαζί με την Eurolat. Και αυτό αποδεικνύει όχι μόνο το ενδιαφέρον, αλλά και την δέσμευσή μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Θα ακούσουμε διάφορους ομιλητές που θα μας παρουσιάσουν την ε, θέση τους για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα. Που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Μιλάμε για καταστολή, συλλήψεις παράνομες, φυλακίσεις, κατάχρηση εξουσίας, πολιτικούς πρόσφυγες, λογοκρισία και ως ανθρωπιστική κρίση που δεν αναγνωρίζει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και ζητάει και δεν ζητάει και απορρίπτει μάλλον τη βοήθεια. Απορρίπτει τη βοήθεια του Μπανκιμού, της Κάριτα και όλων των οργανισμών και φορέων που θέλουν να βοηθήσουν το λαό λόγω τη έλλειψη ε, τροφίμων και βασικών ειδών φαρμάκων κλπ. Αυτό βέβαια θέτει το πληθυσμό σε μια κατάσταση επικίνδυνη. Και γι' αυτό ακριβώ πρέπει να επιθυμίσουμε και την απόρριψη της ε, του αιτήματο επίσκεψη τη Επιτροπή του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόσφατα, σε ψηλό επίπεδο, εκφράσαμε την ανησυχία μας για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αλλά πια έχει έρθει η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Θα θέλαμε να βοηθήσουμε να βοηθήσουμε καταρχάς τους συμπατριώτες μας ως Ευρωπαίοι. Άτομα των οποίων τα δικαιώματα πλήττονται. Καλωσορίζω την Αλεχάνδρα, Αλεχάνδρα Κοσάλες, αδερφή του κ. Κοσάλες, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην φυλακή για πολιτικούς λόγους. Ρωσάωρα Βαλεντίνη επίσης. Ρωσάωρα που είσαι από την Ιταλία σύζυγος του Ζων Κοικοϊτσέα της αντιπολίτευσης που φυλακίστηκε πρόσφατα όπως ξέρετε και στα Κολμενάρες πρώτος ε, φοιτητή που έλαβε άσυλο πολιτικό από την βελική κυβέρνηση. Η Βενεζουέλα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Όχι μόνο επειδή έχουμε αρμοδιότητα για θέματα παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά επειδή άμεσα αφορά συμπατριώτες μας. Αρκετοί κρατούμενοι είναι Ευρωπαίοι. Κάποιοι απεβίωσαν μάλιστα. Άλλοι βρίσκονται σε κάποιες φυλακές σε πολύ κακή κατάσταση. Να χαιρετήσω επίσης και την Μανουέλα Μπολίβαρ, η πρώτη βουλευτής της ε, Βουλής της Βενεζουέλα που επισκέπτεται την Ευρωβουλή. Να σας πω επίσης ότι ο επόμενος προϋπολογισμός δεν πέρασε από την Βουλή της Βενεζουέλας. Παρ' όλα αυτά, σχεδιάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ένα κυρωτικό δημοψήφισμα. Αν γίνουν λοιπόν όλα αυτά, θα φτάσουμε σε κοινωνική ταραχή και χάος ανθρωπιστικό και βεβαίως περαιτέρω παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε να διώξουμε από την εξουσία τον Μαδούρο, αλλά να αντιμετωπίσουμε την κρίση που υπάρχει. Και ξαναλέω, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα νόμιμο μηχανισμό, γιατί έχουμε ένα λαό ο οποίος ανυπόμονα περιμένει την δημοκρατική λύση των προβλημάτων του. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Θα ξανασυζητήσουμε πάντως. Θα θυμάστε ότι τον Ιούνι είχαμε ένα ψήφισμα στην Ευρωβουλή για τη Βενεζουέλα. Η κατάσταση από τότε χειροτέρεψε. Και πρόσφατα στείλαμε μια επιστολή στην κυρία Μογκερίνη. Διάφοροι ευρωβουλευτές ακριβώς για να προειδοποιήσουμε για την κατάσταση που ισχύει. Μετά την επιστολή αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαφίεται στον διάλογο και στη σχέση μεταξύ των τριών πρώην Προέδρων. Αλλά γίνει αυτό, δεν χρειάστηκε να στείλουμε τόσε επιστολέ. Τέλο πάντων, δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Πρέπει να μιλήσουν, πρέπει να μιλήσουν οι προσκεκλημένοι μα. Να θυμίσω ότι στους φακέλους σας έχετε τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε και την Ταμάρα Σούχου από το Ινστιτούτο Κάσλα της Πράγας Πρατρίσια Μπετανκούρ επίσης από τον Μπεν Ευρώπα τώρα μπράβο από την Επιτροπή Θυμάτων της Γουαρίντα και πριν τους δώσω το λόγο σύντομα για τις παρεμβάσεις τους να πω ότι ο κ. Χαουρέγγι, ο πρόεδρος της Ευρωλατ, χρειάστηκε να φύγει, αλλά μας στέλνει μας στέλνει το ενδιαφέρον Συμφωνεί, πολύ απόλυτα επειδή έχουμε καθυστερήσει. Ωραία. 5-6 λεπτά στην καφεμιλήτρια. μιλήτρια. Ας σας παρακαλώ να τηρήσουμε τους χρόνους. Η Ταμάρα Σουκούτ, ναι, η Ταμάρα σε 5 λεπτά μπορεί να τα πει όλα, όλα και παραπάνω. Αλλό, γεια, οκ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω και να σας διηγηθώ τι έχει γίνει του τελευταίους μήνες στην Βενεζουέλα. Είχαμε απειλές, συλλήψεις κατά των αντιφρονούντων και μελών της αντιπολίτευσης το Σεπτέμβριο στην Βενεζουέλα. Η οργάνωσή μας εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της στις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζήτησαν ακυρωτικό δημοψήφισμα. Δημοσιογράφοι διαπομπεύθηκαν με τρόπο κουβανικό. Είχαμε ατιμορρησία ένοπλων ομάδων που τρομοκρατούν τον πληθυσμό και συνεργάζονται με την αστυνομία. Από το Γενάρη του 2014 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 είχαμε 6.536 λήψεις για πολιτικούς λόγους. Για διάφορους λόγους. Αυτή τη στιγμή από τα άτομα αυτά, 101 άτομα, παραμένουν στη φυλακή και χαρακτηρίζονται ως πολιτικοί κρατούμενοι σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. Από την 1η Γενάρη μέχρι 30 Σεπτέμβρη φέτος είχαμε 2.436 συλλήψεις για πολιτικούς λόγους. Από αυτές τις συλλήψεις, τους τελευταίους πέντε μήνες είχαμε 2.219 Κρατήστε το αυτό τον αριθμό. Από τη στιγμή που ξεκίνησε ο υπερθέμενος διάλογος την Πρωτομαγιά στην Βενεζουέλα, είχαμε 2.219 συλλήψεις πολιτικές. 24 έχουν καταδικαστεί και 37 αναμένουν δίκη. 2.055 άτομα που συλλήφθησαν τα τελευταία δύο χρόνια αναμένουν και αυτά τη δίκη. Το καθεστώς λοιπόν της Βενεζουέλας χρησιμοποιεί τις περιστρεφόμενες πόρτες, δηλαδή συλλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, απελευθερώνει, αλλά συνεχίζει να κρατά στη φυλακή. Από τον Ιούλιο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου είχαμε 273 άτομα που συνελήφθησαν και τα οποία διηγηθήκαν στη δικαιοσύνη κρατήθηκαν και 57 απελευθερώθηκαν με περιοριστικούς όρους. Στοιχεία. Γενάρης τρεις συλλήψεις, Φλεβάρι τέσσερις, περνούσε όμως ο καιρός, 100, 200, Ιούνιο 1200 και βάλε άτομα. 900 από αυτά τουλάχιστον συνελήθησαν σε νυχτερινές, βραδινές ουρές μπροστά από σούπερ μάρκετ και φαρμακεία. Σύνολο 2.436 συλλήψεις για πολιτικού λόγους στη Βενεζουέλα. Παρατηρούμε επίσης την καταστολή που αφορά πολιτικού ηθήνοντε τη αντιπολίτευσης. Νέλσον Κοράντα, Γκοϊκοτσέα, Ατάρο, ο δημοσιογράφος, ο Αλεχανδροπύριο, που το μόνο του έγκλημα ήταν να σηκώσει ένα ντρόουν. Έστερ Τολέντο, Βόρνερ Χιμένες, Νταβίτ Μολάσκι. 36 πολιτικοί κρατούμενοι από το Μάη. Είχαμε κακομεταχείριση Επίσης, όπως στην περίπτωση του Μανουέλ Ερνάντες, τον οποίο χτύπησαν ενώ έκανε ουρά, στα κοντά στην ουρά μπροστά από ένα σούπερ μάρκετ. Οι δυνάμεις ε, ασφαλείας δρούν αυθαίρετα όσον αφορά τις συλλήψεις και τις ε, φυλακίσεις και η κακομεταχείριση των πολιτικών κρατωμένων δεν αφορά μόνο την καταπίεση αλλά και την σωματική βία και την απομόνωση απειλές στις οικογένειές τους κάποιοι μάλιστα είχαν εγκλειστεί σε ένα υπόγειο 15 μέτρα κάτω από τη γη μπαίνουν ή τους βάζουν σε απαράδεκτα κελιά χωρίς ιατρική περίθαλψη. Οι συνθήκε λοιπόν αυτές οδηγούν στην υποχώρηση της υγείας τους. Η πλειοψηφία αυτών των ατόμων παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα υγείας, ψυχικής και σωματικής, όπως ο Βλαδιμίρα Ράκε, ο οποίος έχει ένα εγκεφαλικό όγκο και δεν δέχτηκε ιατρική βοήθεια, όπως ο κ. Σορτέγα, ο οποίος έχει φλεβίτιδα και στα δύο πόδια. Ο... Και κρατούμενοι που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Συνεχίστηκαν και τα βασανιστήρια. Ακόμα και την ίδια μέρα που είχαν συναντηθεί οι τρεις ε, πρόεδροι στη Δομικανή Δημοκρατία, συνελήφθησαν 7 νέοι, πήγαν σε αυτή την ε, φυλακή, την υπόγεια, και βασανίστηκαν με ηλεκτροσόκ ή με σεξουαλικά βασανιστήρια, με σακούλες πλαστικές για ασφυξία, όλα αυτά το Μάη. Έχω και άλλα να σας πω, αλλά δεν έχω χρόνο. Ναι, καλά μας τα λες και διεξοδικά, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πάντως, λέει η Πρόεδρος, όπως ξέρετε, οι διερμηνείς καημένοι έχουν και κάποιο ωράριο. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν. Οπότε δεν θα έχουμε διερμηνία να τα πείτε στα αγγλικά. Μπορείτε. Είναι λοιπόν περιορισμένο ο χρόνος. Και εσύ, πέντε λεπτά. Bueno, eh... Γεια σας. Στη Βενεζουέλα διέφυγαν πολλοί Ευρωπαίοι από τον πόλεμο. Η χώρα λοιπόν αναπτύχθηκε με αυτά τα άτομα. Αλλά το φαινόμενο αυτό της μετανάστευσης είναι επίκαιρο, σαν ένα κύμα που γεννιόρχεται ασταμάτητα. Αυτός που πήγε, γύρισε και αυτός που γύρισε, πήγε. Και έχουμε γενιές και απογόνους αυτών των ατόμων που όμως το όνειρο, για τους οποίους το όνειρο έχει γίνει εφιάλτης. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους φυλακισμένους του Μαδουρό. Ευρωπαίους φυλακισμένους που στο πετσί τους νιώθουν ακριβώς την βία και τις αφαιρεσίες που μας ανέφερε προηγουμένως η Ταμάρα, οι η οι Πορτογάλοι, οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα στη χώρα και οι οποίοι ξεχάστηκαν από τις πρεσβείες και τα προξενία τους. Ο κατάλογος που παρουσιάζουμε συντάχθηκε με μεγάλες δυσκολίες με τη βοήθεια μιας ένωσης για τα δικαιώματα που προσπάθησε ή προσπαθεί να βοηθήσει τους κρατούμενους σε όλα τα επίπεδα. Γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να ανακαλύψει καλή τους Ευρωπαίους, γιατί είναι ταυτόχρονα και υπήκοοι Βενεζουέλα. Και επειδή τα επώνυμά του καμιά φορά δεν είναι διαφορετικά, περνάνε απαρατήρητοι. Θα θέλαμε λοιπόν να καταγγείλουμε περιπτώσεις δεκάδων ατόμων που έχουν καταναμηθεί σε διάφορες φυλακές και που έχουν υποστεί τις ίδιες απάνθρωπες συνθήκες και αυθαιρεσίες. Δεν έχω χρόνο, αλλά να σας πω τα ονόματά τους και τις εθνικότητες τους. Μας ανέφερε ήταν παραπηγουμένως σε τι υπόκεινται. Τα ονόματα τους είναι. Βρέου, Πορτουγές. Μπέτι Γρόσι, Ιταλιάνα. Βάσκο Δακώστα, Πορτουγές. Alejandro Pulla, italiano. Iván Simonovis, español. Andrés Thompson, inglés. Raúl Emilio, Emilio Baduel Cafarelli, italiano. Josefa de González, española. Ignacio Porras, español. Αυτά ήταν τα ονόματα και εθνικότητες. Είναι Ευρωπαίοι αυτοί, ταπεινωμένοι και καθένας από αυτούς εκπροσωπούν την Ευρώπη, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Εντάξει, βρίσκονται σε μια απόσταση χιλιάδων χιλιόμετρων, αλλά αυτό δεν τους καθιστά πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Γι' αυτό θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε ό,τι μπορείτε, ώστε καταρχάς να μάθουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτοί οι Ευρωπαίοι. Να πιέσουμε ώστε τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Καράκας να τους επισκεφτούν και να ζητήσουμε να υπάρξει περιβόητη αποστολή της Ευρωβουλής στη Βενεζουέλα και να περιλάβει στις επισκέψεις που θα κάνει και αυτούς τους Ευρωπαίους. Μέχρι πού φτάνουν λοιπόν τα σύνορα της Ευρώπης, τα σύνορα των αρχών και των αξιών της. Κάθε πολίτης είναι από μόνος του ένα σύνορο της χώρας του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πατρίθια. Στην κυρία Σωρέτα, μπράβο, θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα για πέντε λεπτά. Γεια σας. Με λένε Σωρέτα, μπράβο από την Επιτροπή Θυμάτων της Γουαρίμπα, μια μη κυβερνητική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορά θύματα και συγγενείς θυμάτων πολιτικής βίας που έλαβαν χώρα στη Μεζουέλα το 2013 και το 2014. Με συνοδεύει ο κύριος Οσκαρ Καρέρο, μέλος και αυτός της Επιτροπής μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την υποπιτροπή σας για την πρόσκληση. Φέτος τηρήσαμε ενήμερο το Κοινοβούλιο και τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς σχετικά με τα θύματα της βίας στην χώρα μας. Πέρσι συναντηθήκαμε μια αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής που ήρθε στο Καράκας και πρόσφατα συναντήσαμε την Γενική Διευθύντρια για τη Λατινική Αμερική της ΕΙΕΔ. Δεν αρκούν βέβαια όλα αυτά για να γνωστοποιήσουμε την καταπίεση και τη θανάτωση των συγγενών μας και να ζητήσουμε δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο γιος μου. Αυτός είναι ο γιος μου. Λοχαγός μπράβο. Τον δολοφόνησαν το Μάρτιο του 14 ένας μήνες δολοφονίας έχουν περάσει. Όταν λοιπόν ομάδες ενόπλων προσπάθησαν να κάψουν ένα βενζινάδικο, είχαμε καταγγελία και προσπαθήσαμε να πάμε, αλλά μας περίμεναν ένοπλες δυνάμεις αυτές οι βίαιες ένοπλες δυνάμεις πυροβολούσαν τους στρατιωτικούς που προσπαθούσαν να προστατεύσουν τον πληθυσμό. Προσπάθησε ο γιος μου να προστατεύσει έναν τραυματία, αλλά μια δέσποτη σφαίρα τον σκότωσε. είχαμε πάνω από 43 νεκρούς και 800 τραυματίες. Σας έχουμε φέρει πληροφορίες για όλα αυτά τα συμβάντα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ώστε η ηλική και η ηθική υπεύθυνη για αυτά τα συμβάντα να καταδικαστούν ώστε να μην ξανασυμβούν αυτά τα γεγονότα στη χώρα μας. Να σας πω ότι για μας θα είναι πολύ δύσκολο να ξανάρθουμε γιατί έχουμε την εντύπωση ότι δεν μας προστάτευσε αρκετά το κοινοβουλίο σας ως θύματα στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. και οι υπεύθυνοι αυτών των εγκλημάτων έμειναν ατιμόρυτοι. Πάντως, θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη των συγγενών μας που θανατώθηκαν λόγω των, λόγω των ακραίων στοιχείων της κοινωνίας της Βενεζουέλας. Η αλήθεια, κυρίε και κύριοι βουλευτές, είναι ότι η οργάνωσή μας θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε να μην υπάρχει ατιμορρυσία. Υποστηρίξαμε την δημιουργία της Επιτροπής Αλήθειας, ώστε να εξεταστούν σε βάθος όλες οι υποθέσεις αυτές και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση και θα θέλαμε να ζητήσουμε από τα μέλη του Κοινοβουλίου σας να κάνουν τα απαραίτητα ώστε να σταματήσει η βία που προκάλεσε τόσους θανάτους. Διεκδικούμε το δικαίωμα για ειρηνικέ διαδηλώσεις χωρίς βία. Ο αγώνας μας αποβλέπει στο να διελευκανθούν οι περιστάσεις στις οποίες συμμετείχαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης και συμβάτα τα οποία δείξαν σε θάνατο αθών. Το κοινοβούλιο σας πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά της οργάνωσής μας. Θα θέλαμε να ζητήσουμε να μην, υπάρχει, να μην υπάρξει ατιμορρησία των θητών και ζητάμε με, για όλα τα θύματα αυτών των δράσεων. Θα θέλαμε επίσης να σας ζητήσουμε να στηρίξετε τη συγκρότηση της Επιτροπής Αληθείας για την διαλεύκανση όλων των συμβάντων και την αναζήτηση των υπευθύνων που προκάλεσαν το θάνατο 43 ατόμων και τον τραυματισμό πάνω από 800. Θα θέλαμε το Κοινοβούλιο να στηρίξει τη δικασία διαλόγου στη Βενεζουέλα. Μέσω και της πρωτοβουλίας των τριών πρόεδρων. Και καλούμε όλους τους τομείς της κοινωνίας της Βενεζουέλας να μην χρησιμοποιήσουν τη βία για πολιτικούς λόγους. Θέλουμε να κρατήσει ο διάλογος. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ κυρία Μπράβο. Ζήσαν το λόγο διάφοροι συνάδελφοι. Να σας πω τη σειρά λόγου. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Γιατί πάνω από ένα λεπτό θα είναι δύσκολο. Σενιόρ Λουίς Δε Γκράντες. Λουίς Δε Γκράντες, Καταρχάς. Και μετά κύριο Σταγιάννη. Ταγιάννη, Ροντρίγες, Φαρία, Κόουσο, Χιμένες Μπεθερίλ. De Grandes. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμμερίζομαι όλα σας τα λόγια. Η διάγνωσή σας μάλιστα συνοδεύεται και από αυτά που είπαν οι προσκεκλημένοι μας. Θεωρούμε ότι ο αυτοχειρισμός του καθεστώτος Μαδούρο έχει οδηγήσει σε άνευ ορίων καταστολή. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε στρατιωτικούς, σαν να ήταν σκέδους κυβέρνηση, ήταν, είναι κάτι αντιδημοκρατικό. Και συνεχίζεται ο εκφαβισμός και η τρομοκράτηση του λαού της Βενεζουέλας. Κυρία Πρόεδρε, έτοιμα. Να ζητήσουμε επισήμως από την πρέσβυρα της Βενεζουέλας να έρθει εδώ ιδιαίτερα σε σχέση με τον κύριο Γιόν Κοεκοετσέα, ένα κρατούμενο, για να μάθουμε ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται και πώς θα μπορούσε κανείς να προστατεύσει ένα θαραλέο ηγέτη, ο οποίο βρίσκεται στη φυλακή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σταγιάννη. Παραμένει δραματική κατάσταση στην Βενεζουέλα. Λείπουν φάρμακα. Έχουμε διακοπή των προγραμμάτων εμβολιασμού, κάτι το οποίο προκαλεί θανάτους. Έχουν αυξηθεί και λόγω διφθερίας θάνατοι βρεφών. με παιδιά τα οποία βρίσκονται νεκρά σε κουτιά. Είναι απίστευτο αυτό. Έχουμε πληθωρισμό 1600% σχέση με το τωρινό 400%. Πριν λίγους μήνες είδαμε κόσμο να ζητιανεύει για φαγητό στον δρόμο. Υπάρχει μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν πολλά εμεί, όπω είπαν και οι συνάδελφοι, να καλέσουμε εδώ την πρέσβυρα να μα πει τι γίνεται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Βενεζουαλανών. Ο Μαδούρο για μένα είναι δικτάτορα. Πρέπει όμω να προσπιστούμε τα δικαιώματα των μωρών, των γυναικών. Βλέπετε τι γίνεται καθημερινά. Έχουμε μια κατάσταση που είναι καταστροφή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν να ζητήσουμε από την πρεσβεία και την πρέσβυρα να μας πει τι κάνει η κυβέρνησή τους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και βεβαίω πρέπει να έχουμε και μια αποστολή. Να σας ενημερώσω επίσης ότι η μεικτή συνέλευση με την Ευρωλάτ ψήφισε πριν δύο εβδομάδες μια έκθεση όπου γίνεται λόγο ξεκάθαρα για την επικίνδυνη κατάσταση στη Βενεσουέλα. Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση αυτή είναι επικίνδυνη για όλους, κυρίως για την Ευρώπη, γιατί έχουμε και πολιτικούς κρατουμένου Ευρωπαίους. Έχουμε πολλούς Ιταλούς, σαν και εμένα, που ζουν εκεί και έχουμε σοβαρές ανησυχίες για τους Ιταλούς και για τους Βενεζουαλούς Ιταλικής καταγωγής. Ευχαριστώ, αλλά φοβάμαι θα μείνουμε χωρίς ε, διερμηνία, γιατί ζητήσαμε περισσότερο χρόνο από ό,τι μπορούμε. Σημειώσαμε πάντως τα αιτήματά σας. De Venezuela, por supuesto, ha sido eh, invitada hoy, como en anteriores ocasiones,